Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το τμήμα της κοινής συνεδρίασης Μπουτζέκον. Ε, Έχουμε μόνο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι η δημιουργία της ε, ευρωπαϊκής λειτουργίας ε, σταθεροποίησης των επενδύσεων. Να ξεκινήσουμε τους συζητητές. Έχουμε γύρω στα 40 λεπτά αυτή τη συνεδρίαση. Λοιπόν, αρχίσουμε με την Περβάς Μπερές που είναι η συγήτρια ε, από πλευράς έκον των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που οι δύο επιτροπές μας ε, έχουν αυτή τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις για τις τροπολογίες που υπευλήθησαν. Είναι πάνω από 400 οι συνεισηγητές υποβάλαμε και εμείς κάποιες. Να σας εξηγήσω την προσέγγιση με βάση την οποία ε, ο κύριος Μπέγκη και εγώ τροποποιήσαμε το σχέδιο εκθεσής μας μετά τις, ε, συζητήσεις που έγιναν κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο εκθεσής μας και μετά τις επαφές που είχαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά αλλά και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαν οι απόψεις μας από αυτά τα οποία είπε στη γνωμοδότησή της και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από κάποιες εργασίες που διεξάγονται τώρα στο Συμβούλιο. Γι' αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να διευρύνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θυμάστε ότι είναι μια πρόταση που υπό ορισμένε προϋποθέσεις προτείνει εάν ένα κράτος μέλος με βάση κάποια κριτήρια αντιμετωπίζει προβλήματα ανεργίας να δημιουργηθεί ένας αυτόματος μηχανισμός σταθεροποίηση, όπως λέει και το όνομά του η πρόταση της Επιτροπής λέει ότι αυτή η σταθεροποίηση θα γίνεται μέσω στήριξης των επενδύσεων εμείς προτείνουμε να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα αλλά να συμπληρωθεί με τη δυνατότητα παρέμβασης όχι μόνο στον τομέα της προσφοράς αλλά και τις ζήτησης ε, για αυτή την αυτόματη σταθεροποιητική προσπάθεια, στηρίζοντας τα εθνικά συστήματα επιδομάτων ανεργίας. Να υπάρχει ένα είδος αντασφάλισης. Δεν παρεμβαίνει με τις διατάξεις, στις διατάξεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη για τις ε, σχέσεις των κοινωνικών εταίρων, αλλά μπορεί όντως να ε, επηρεάσει θετικά εντόνως ε, αυτή την προσπάθεια σταθροποίησης. Αυτά θέλω να πω εγώ. Θα συμπληρώσει και ο Ράινερ Μπέγκε. Νομίζω ότι είναι επίγουσα αυτή η πρόταση. Γιατί βλέπουμε τι συζητήσει γίνονται στο Συμβούλιο και μα ανησυχούν κάπω. Γιατί αυτό ο στόχο που έχει εντοπιστεί από όλου και τον αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι απαράδεκτο για να υπάρξει βιωσιμότητα τη ζώνη ευρώ, δεν αντιμετωπίζεται ουσιοδό σε διάφορε άλλε εργασίε αλλού. Αυτοί που θεωρούν ότι τις επόμενες κρίσεις ε, μπορεί να ασφαλιστοποιηθεί ή κρίσεις μπορεί να τι αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη χωρίς αυτή τη ε, λειτουργία σταθεροποίηση, τις απόψει αυτές δεν τι θεωρώ ε, βάσιμες. Αυτά κοίταξα μαζί με τον Ράινερ όλες τις τροπολογίες. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που θεωρούμε απόλυτα χρήσιμες, αλλά... Κοιτάξτε, Είμαστε σε αυτή τη ε, φάση της ε, θητείας και πρέπει να συμφωνήσουμε συνάδελφοι μεταξύ του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών. Θεωρούμε ότι ε, εφόσον έχουμε συμφωνήσει εμεί αυτή τη βάση, θα πρέπει να είναι η βάση από τι οποίε θα πρέπει να καθορίζουν τη στάση τους και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρο, και ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο ομιλία σα, τον οποίο ούτε καν ανέφερα όμω. Τέσσερα λεπτά. Οπότε όμω τέσσερα για τον κύριο Μπέγκε. Το πολύ προ, ε, κύριε Μπέγκε, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κύριο Μπέγκε. Σημείο αφετηρία ημών των συνεισηγητών ήταν αυτά που συζητήσαμε τον Φεβρουάριο του 2017 σε μια πρόταση πρωτοβουλία, έκθεση πρωτοβουλία που πέρασε από την Ολομέλεια, που μπορεί να δημιούργησε κάποιε διαφωνίε, αλλά πέρασε με ευρία πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Πέρασε τώρα, περάσαμε τώρα στη φάση μια νομοθετική πρόταση τη Κομισιόν. Νομίζω ότι ο οποίος ε, εκφράζεται για αυτά τα διάφορα μέσα και αυτό είναι και το αίτημά μου πρέπει να έχει καταλάβει σαφώς ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα με την πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που παράλληλα προβλέπει μια σειρά ε, επεκτάσεων των υπαρχόντων δυνατοτήτων αλλά προτείνει και ορισμένες νέες δυνατότητες και αυτό είναι μάλλον ένα τμήμα του προβλήματος δεν έχει να κάνει με τη δική μας ε, έκθεση και αυτό το μηχανισμό σταθεροποίησης των επενδύσεων, αλλά γενικά ότι πρέπει να έχουμε μια ε, συνεκτική ε, συνολική προσπάθεια. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε όπως το συζητήσαμε και στην συνεδρίασή μας των σκιωδών την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Έχουμε την πολιτική συνοχή, έχουμε το κοινωνικό ταμείο, έχουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου πώς πρέπει να διαμορφωθούν αυτά στο μέλλον, πού πρέπει να έχουμε επιπλέον δυνατότητες. Έχουμε το InvestEU, που είναι η συνέχιση του προγράμματος Juncker, και έχουμε και την πρόταση της κυρίας Γαρδιαθάβαλ, πώς όλα αυτά συνδυάζονται, ώστε να αποτελούν ένα σύστημα. Ε, θα πρέπει να υπάρχει άμεση, κεντρική διαχείριση, ε, μοιρασμένη διαχείριση. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά ε, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πού εντάσσεται η δική μας έκθεση σε όλα αυτά. Πολλοί και τους ε, καταλαβαίνω λένε ότι πρέπει να συζητηθούν μαζί όλα αυτά τα μέσα, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί για να έχουν έννοια. Και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι και εγώ ως Κάτι άλλο. Είδαμε ότι έχουμε πάνω από 400 τροπολογίες. Εκφράζουν πολύ διαφορετικές απόψεις, αυτό είναι αναπόφευκτο. Άλλοι υποστηρίζουν και περαιτέρω αναπτύσσουν την πρόταση της Επιτροπής, ενώ άλλοι υποβάλλουν τόσο περίπλοκες τροπολογίες που δεν είναι δυνατόν να τις ε, δεχθώ. Πρέπει να σας τα πω τα πράγματα όπως είναι. Θέλω λοιπόν να τονίσω Χωρί να πω ότι τα καταλαβαίνω όλα και έχω πλήρη άποψη για όλα, ότι εάν η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας συμβαδίζει με την πρόταση της Κομισιόν, εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι το συζητήσαμε και σε μια βίντεο σύνδεση, όταν είχαμε τότε την έκθεση πρωτοβουλίας. Εάν έχουμε μια πρωτοβουλία 14 ειδικών Γάλλων και Γερμανών ε, που συμφωνούν με αυτή την κατεύθυνση κάνοντας κάποιες ε, συμπληρώσεις νομίζω ότι πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά πολύ σοβαρά και να τα δούμε πολύ συγκεκριμένα για μένα δύο αποφασιστικά που θα υπάρξουν και στις ε, κοινέ τροπολογίες που υπήρχαν και στην έκθεση πρωτοβουλίας πρώτα απ' όλα να έχουμε ένα σύστημα ασφάλισης πώς θα διαμορφωθεί ούτως ώστε ο καθένα ε, με σαφεί συνθήκε ε, να έχει ε, πρόσβαση σε ορισμένα επιδόματα και να είναι και επίσης δημοσιονομικά ουδέτερο μακροπρόθεσμα. Αυτά είναι τα αποφασιστικά. Και οι συνάδελφοι που έχουν κάποιες δυσχέρειες με αυτή την διατύπωση σύστημα αντασφάλισης και ασφάλιση των επενδύσεων να δείτε το αρχικό ε, άρθρο 5 που δεν το θίγουμε εμείς. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να εγγυόμεθα κάποιες επενδύσεις κάποιου επίπεδου και αν δεν γίνεται αυτό τότε να παρενεβαίνει η Κομισιόν. Αυτό είναι το τμήμα του συστήματος το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε. Η πρότασή μας τελικά είναι μια προσπάθεια να κάνουμε μια δεύτερη συνεδρίαση των σκιωδών πριν ε, τα Χριστούγεννα για να καταλήξουμε σε ένα πακέτο που δεν θα μπορέσει ωστόσο να ψηφιστεί σε μια κοινή ε, συνεδρίαση των δύο επιτροπών τον ε, Δεκέμβριο, αλλά να το συζητήσουν οι πολιτικές ομάδες τον Δεκέμβριο και να το αποφασίσουν τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ κύριε Μπέγκη. Χρησιμοποιήσατε και το λεπτό που άφησε η συνεισηγήτρια. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ορίσατε το πλαίσιο της συζήτησης. Περνάμε τώρα στους οι εισηγητές. Ξεκινάμε με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και τον κύριο Ντό Σάντος από τους Σοσιαλιστές. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η εκθέση αυτή ε, έχει περιγραφεί σωστά από τους συνεισηγητές. Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντική αφορά δύο ζητήματα που συζητούν οι επιτροπές μας και η γενική μου θέση είναι ότι συμφωνώ σε γενικές γραμμές με την πρόταση και την ε, προσέγγιση της Περβάνς Μπερές. Παρ' αυτά, έχω κάποια ζητήματα μεθοδολογίας όσον αφορά τον ορισμό των στόχων της έκθεσης, αντιλαμβάνομαι την προσέγγιση της Περβάνος Μπερές και το κίνητρο των τροπολογιών της ε, στηρίζω και έχω συνυπογράψει πολλές ε, στις Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού αλλά εδώ πέρα έχουμε πολύ περίπλοκα ζητήματα και σε πολλές ε, περιπτώσεις δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε αξιολογικές ε, συμβαστικές ε, προτάσεις. Γι' αυτό και αναβλήθηκε η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι αναδεικνύεται η ανάγκη να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της έκθεσης. Έχω υποβάλει και εγώ κάποιες ε, τροπολογίες. Όπως είπα, συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ΕΚΟΝ Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού οι τροπολογισμοί αφορούσαν ε, τρία κυρίως πράγματα. Το πρώτο ήταν τα κριτήρια για πρόσβαση στο Ταμείο, δηλαδή την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο, αν και σε πολλές περιπτώσεις βεβαίω ε, συμπίπτουν. Δεύτερον, υπάρχει η δυνατότητα, η το μέγεθος δηλαδή του ταμείου που πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Μιλάμε για ένα επίπεδο χρηματοδότησης που θα πηγαίνει πολύ πέρα από την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Και μέσω των τροπολογιών που έχω υποβάλει ε, λέω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στις χώρες της Ευρωζώνης ε, και τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Αυτές είναι οι τροπολογίες μου. Και ε, πρέπει να πω ότι υποστηρίζω τις περισσότερες ε, από αυτές που προτάθηκαν στην ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μούρεσαν από την Επιτροπή Οικονομικών και το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω να προεδρεύετε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περβάνς και τον Ράιμερ Μπέγκε για το σχέδιο έκθεσης που υπέβαλαν. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο θέμα στο οποίο οι απόψει αποκλίνουν, γι' αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που το επέβαλαν και προσπαθούν να συμβιβάσουν τις απόψεις. Βεβαίως υπάρχουν πολλές τροπολογίες από διαφορετικές πολιτικές ομάδες και την δική μου. Εγώ είμαι σκιώδης ε, συγητής ε, του ΕΛΚ ε, στην Έκονο. Συντονιστής μας έχει υποβαλεί 20 τροπολογίες νομίζω. Λοιπόν, τι θέλουμε εμείς ως ΕΛΚ βεβαίως συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και καθώς ε, σκεφτόμαστε την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού ενός Ζατικού Ταμείου θα πρέπει ακριβώ να έχουμε τα σωστά κίνητρα και όρους ένα μέσο δηλαδή το οποίο θα βοηθάει τις χώρες που έχουν δυσκολίες γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ορθή συμπεριφορά όσον αφορά την ε, συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ε, την ενθάνση των μεταρρυθμίσεων. Και πριν ε, μπουν σε μια κρίση και βεβαίως δεν θα πρέπει να έχει μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος η χώρα πριν γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τις χώρες εκείνες οι οποίες διαχειρίζονταν σωστά τα δημόσια οικονομικά τους και τα πλήτη μια αναπάντεχη κρίση. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι ο ξεκάθαρος ορισμός των ασύμμετρων κραδασμών είναι κάτι το απαραίτητο. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ορισμός και βεβαίως έχουμε προτείνει τον περιορισμό των χωρών ε, στο 1 τρίτο γιατί αν μιλάμε για πάνω από το 1 τρίτο των χωρών δεν μιλάμε για ασύμμετρο κραδασμό πλέον αλλά για συμμετρικότατο. Και βεβαίω ε, το κρεμές ποσό των δανείων θα πρέπει να είναι περιορισμένο και η χορήγηση δανείου θα πρέπει να είναι ανάλογα με την διαθεσιμότητα που υπάρχει όσον αφορά το σχέδιο αυτό της αντασφάλισης ανεργίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι κόκκινη γραμμή για πολλούς συναδέλφους Οπότε αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση εντός της ομάδας και εντός του Κοινοβουλίου και για να καταλήξω κύριε Πρόεδρε. Για να επηρεάσουμε το Συμβούλιο στο θέμα αυτό χρειάζεται μια ξεκάθαρη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Όταν εγκρίναμε την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας είχαμε 304 ψήφους υπέρ, 255 κατά και 68 αποχές. Τώρα λοιπόν σοβαρά τα πράγματα είναι συνομοθεσία πρέπει να επηρεάσουμε το Συμβούλιο πρέπει λοιπόν να είμαστε ενωμένοι με μια σαφή πλειοψηφία για να έχουν και ισχυρή εντολή οι Σε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μανσάν. Σοφά τα λόγια σας. Να σας θυμίσω ότι θέλω να τηρείτε το δίλεπτο στις παραβάσεις. Ότως ώστε η ροή να είναι καλή στη συζήτηση για δύο λεπτά. Ο κ. Κέλμερ, που είναι εισηγητή του ECR για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι οι εισηγητέ, οι συνεισηγητέ, ήσαν ιδιαίτερα επιμελεί. Και χθε όμως που συζητούσαμε ένα περαιτέρω μέτρο, είμαι 100% ο σίγουρος ότι είναι λάθος αυτή η πορεία. Αυτά τα μέτρα μας αποπροσανατολίζουν από το βασικό πρόβλημα. Τακτικά λέμε εδώ ότι το ευρώ είναι επιτυχημένο, ότι τα πάμε καλά, αλλά στην πράξη κάθε δύο μήνες ε, γεννιούνται νέα όργανα, νέοι μηχανισμοί και λέμε βεβαίως το χρειαζόμαστε και αυτό. Και αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι θελημένα γίνεται κατάχρηση της λέξης ε, αλληλεγγύη. Είναι σημαντική αλληλεγγύη και υπάρχει στην Ένωση. Όμω, αν μια χώρα, επειδή έχει διευθυντικά προβλήματα, δεν είναι σε θέση να πληρώνει του λογαριασμού τη και να διατηρεί ένα ε, τραπεζικό σύστημα που να λειτουργεί, τότε πια δεν είναι θέμα αλληλεγγύη, Εάν αυτοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν την οικονομία του ή εάν ε, είναι σπάταλοι. Κάθε χώρα πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της και να πληρώνει ε, όσα καταναλώνει. Με τέτοια μέτρα τα οποία εισάγουμε τώρα, τότε τα κάνουμε όλα φλού. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Αυτό είναι φταίνουν όλοι για όλα. Ο καθένας κάνει τη γουστάρει και το αποτέλεσμα υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Είμαι κάθετα εναντίον τέτοιων μέτρων όπως είπα επανελειμμένα, είναι απόλυτα αδιαφανή. Αν δούμε τι μέτρα έχει λάβει το μεταξύ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε η πολιτική των μηδενικών επιτοκίων τουλάχιστον έχει κάποια διαφάνεια. Όμως ε, τώρα αγοράζουν και τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα οι ε, δικαιωμένες εφημερίδες, ναι, ναι, τελειώνω, ότι σκέφτονται να διασώσουν πάλι το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα με ένα ειδικό μέσο. Μα καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Από διάφορα ε, τσουκάλια βουτάμε εκατοντάδες και να, θα πληρώσω το λογαριασμό σε επόμενες εκλογές. Ευχαριστώ κύριος Λούκε. Η Κονίσια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπέγκε τόνισε πως 14 Γάλλοι και Γερμανοί επιστήμονες έχουν στήριξει την πρόταση αυτή. Βεβαίως πρέπει να τα δούμε αυτά στο σωστό πλαίσιο. Δηλαδή στην Γερμανία υπάρχουν γύρω στους 600 καθηγητές οικονομικών και φαντάζομαι ανάλογος θα είναι και ο αριθμός στην Γαλλία. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε για ποιον λόγο 1500 καθηγητές δεν ακολούθησαν αυτούς τους 14. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι η πρόταση αυτή είναι λανθασμένη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λανθασμένη από την ρίζα της γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη νομική βάση και πρόκειται πράγματι για μια προσπάθεια της ε, Κομισιόν να δράσει ούλτρα εκτός δηλαδή των αρμοδιοτήτων της ε, Μιλάμε για τα άρθρα 164 και 165 τα οποία αναζητούνται ως νομική βάση, την πολιτική συνοχή. Αυτό όμως το οποίο συζητάμε εδώ πέρα δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική συνοχή. Προτείνεται η προώθηση δημοσίων επενδύσεων σε μια χώρα η οποία έχει πληγεί από υψηλή ανεργία και δεν αναφέρεται πουθενά ότι θα βοηθηθούν οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές μιας χώρας. Άρα ούτε μία σχέση με πολιτική συνοχή επιπλέον κάθε χώρα της Ευρωζώνης ε, και στον, ε, που συμμετέχει στο δεύτερο μηχανισμό συναλλαγματικών ε, ισοτιμιών μπορεί να προσφύγει σε αυτό το μηχανισμό και χωρίς ε, τόκους ακόμα και το Λουξεμβούργο μάλιστα. Δηλαδή τι σχέση έχει το Λουξεμβούργο με μειονεκτική περιοχή που διασφαλίζουμε ότι το μέσο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για μειονεκτικές περιοχές όταν κάθε χώρα της Ευρωζώνης μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Οπότε η παράκλησή μου προς εσάς κύριε Πρόεδρε και στον Πρόεδρο της ΕΚΟΝ ο οποίος δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή είναι να ζητήσουμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας ε, του Κοινοβουλίου. Εδώ πέρα δρούμε ουλτραβύρης και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό πριν βρεθούμε in medias res όσον αφορά τους οικονομικούς μηχανισμούς. Ε, πρέπει να το δούμε αυτό νόμικα πριν ε, προχωρήσουμε και εγκρίνουμε μια τέτοια πρόταση νόμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. 7 δευτερόλεπτα λιγότερα από τον συνάδελφό σας του ECR και ένα λεπτό λιγότερο από ό,τι οι συγητές του ΕΛ και των σοσιαλιστών, αν επιτρέπετε, Πρόεδρε. Λοιπόν, σκέδος υπολογισμού για την ΑΛΤΑ ο κ. Πάιτ δεν παρίσταται δυστυχώς. Σκιώδης τη Ίκων από Λουασάντα. Ο κύριο Τρεμό, εμπάρ σας, Θα προσπαθήσω να μιλήσω για ένα δίλεπτο. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στους εισηγητέ. Από τις συνάδελφοι χτε στην ίδια αίθουσα είχαμε τον Μάριο Ντράγκη. Αναφάθηκε στην ε, ευρωπαϊκή προσπάθεια ε, για την σταθεροποίηση ε, της Ευρωζώνης. Ξέρετε ότι η ομάδα των φιλελευθέρων ήταν πάντα ευαίσθητη για αυτά τα ζητήματα, για την αιρεσιμότητα, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τους ε, κανόνες που έχουμε θεσπίσει για την οικονομική διακυβέρνηση. Νόμους που ψηφίσαμε πρόσφατα και ο Μάριο Ντράγκη χθε αναφέρθηκε στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ χωρών για συμμόρφωση με τους κανένες και την επίτευξη συγκλήσεως. Αυτού του είδους τα βήματα προσπαθούμε να πετύχουμε σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην Ευρώπη θα ήταν πολύ ευκολότερα αν είχαμε άλλε συνθήκε. Ποια είναι η πραγματικότητα σαν φιλελεύθεροι κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες σε κάποια κατημέλη που διαπιστώνουν τα τελευταία χρόνια. Αν υπάρχει ασύμετρο κλειδονισμό, μπορεί να έχει σημαντικό δραματικό αντίκτυπο στις δημόσιες επενδύσεις. Άρα χρειαζόμαστε μέσα, εργαλεία, να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο. Οι φιλελεύθεροι θα υποστήριζαν αυτόματες επενδύσεις, αλλά με ρησιμότητα. Ναι, τα, τα προγράμματα να αφορούν δημόσιε επενδύσεις χωρίς αιρεσιμότητα όσον αφορά τα μακροοικονομικά ε, αποτελέσματα, μακροοικονομικό αντίκτυπο. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε επικοινωνικές συνθήκε κατασκευάζοντας αεροδρόμια χωρί αεροπλάνα και αυτοκινητόδρομους χωρίς ε, κυκλοφορία. Είμαστε ευαίσθητοι όσον αφορά την αυτόματη αντασφάλιση για την ανεργία σαν μηχανισμό να βοηθήσουμε χώρες που έχουν υποστεί ασύμετρο κλειδονισμό σε αυτή την ένωση όπου υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις στην κρίση. Γι' αυτό θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα. Ευχαριστώ. Πράσινη. Ο κ. Σολέ, που είναι σκιώδης ηγετής για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές πρώτα απ' όλα για το έργο τους. Υποβάλαμε αρκετές τροπολογίες. Συμφωνούμε με τη λογική της προτάσεως. Θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Χρειάζονται όμως κάποιες βελτιώσεις. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία. Πρώτα απ' όλα το μέγεθος είναι πολύ μετριοπαθές της προτάσεως θέλουμε να ανέλθει τουλάχιστον στο 1% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Άρα διπλάσιο από αυτό που προτείνουν οι συνεισηγητές. Στην τροπολογία 19 για την ερεσιμότητα θα πρέπει εκεί να συμπεριληφθεί κάποια μορφή κοινωνικών περιβαλλοντικών ε, παραγόντων πέρα από τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Φερρυπίν συμμόρφωση με ενδιάμεσους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσης για το 2020 και για τη διάδραση μεταξύ λειτουργίας σταθεροποίησεως και ε, το διάδοχο του ESM, οι τροπολογίες 26 και 27 των συνεισηγητών διαγράφουν διατάξεις που επιτρέπουν συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων. Διαφωνούμε με τέτοιες διαγραφές. Πιστεύουμε ότι τέτοιες διατάξεις θα επέτρεπαν στο μέλλον ενδεχομένως αύξηση ευέλικτη της λειτουργίας σταθεροποίησεως που είναι πολύ μετριοπαθής στην πρόταση και αυτό θα μπορούσε να είναι συμπροματικό μέτρο όσον αφορά το κοινοτικό οι ιδεώδες για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και νομίζουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η αλληλεξάρτηση, αυτή η διάδραση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την εικόνα και ο Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στον ε, κύριο Μπέγκε ότι όταν λέτε ότι αυτό πρέπει να το δούμε μαζί με το InvestEU να σας υπενθυμίσω ότι το λεγόμενο σχέδιο Juncker έχει καταλήξει σε πολλές επενδύσεις σε χώρες όπως η δική σας όπου ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές επενδύσεις οπότε έχουμε προφανώς ένα πρόβλημα στόχευσης το πρόβλημα δεν είναι στη Γερμανία ή στο Βέλγιο εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα επενδύσεων είναι μάλλον σε χώρες όπου δεν υπάρχει ε, πρέπει να το έχουμε αυτό κατά και αν δείτε την στόχευση του πράγματος κάναμε εδώ πέρα μία προσωμείωση και βεβαίως ε, θα έπρεπε να έχει αδρανοποιηθεί το 2014 οπότε, ενώ ξέρουμε ότι χρειάζονται ακόμα επενδύσεις οπότε όσον αφορά τα κριτήρια πρώτο αναρωτιόμαστε πως θα έπρεπε να επιβάλλουμε την ε, ταυτόχρονη πλήρωση των δύο σωρευτικών όρων και θα, θα πρέπει να πούμε όχι αν θέλουμε περισσότερη στόχευση και να εξαιρεθούν τουλάχιστον τα κράτη-μέλη που έχουν ε, ανεργία πάνω από το μεσόρο της Ευρωζώνης από το να πληρώνουν τους δύο όρους ε, ταυτόχρονα. Όσον αφορά τις εθνικές ε, συνεισφορές και η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν ως ε, κριτήριο, το, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το εάν πληρούνται τα ζητήματα που αφορούν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες γιατί κάποιες χώρες βεβαίως έχουν μια μακροοικονομική πολιτική που βλάπτει άλλες και πρέπει να κινηθούν αναλόγως δηλαδή αν βλάπτει ε, η μακροοικονομική πολιτική τους θα πρέπει να χρηματοδοτούν αυτό το ταμείο που ακριβώς αντισταθμίζει τον αρνητικό αντίκτυπο των πολιτικών τους και βεβαίως ε, για τον τύπο των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να στοχεύουμε σε επενδύσεις έτσι ώστε να μας βοηθούν να πολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτς. Η Γκουε. Μετά. Είναι εδώ πέρα κάποιος. Όχι. Κανείς τους δεν είναι εδώ. Πάμε παρακάτω. Η FTD. Ο βάλει είναι εδώ. Όχι, κανένας Μάρκος δεν είναι εδώ. Η ΕΝΕΦ ούτε εκεί πέρα κανένας Μάρκος. Οπότε ένας βουλευτής έχει ζητήσει τον λόγο. Η κυρία Ροντρίγκε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω ότι βλέπω ότι η δουλειά της κυρίας Μπερές και του κυρίου Μπέκε είναι πολύ χρήσιμη και επικοδομητική. Είναι πολύ σημαντικό να δραστηριοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όταν υπάρχει μια σειρά αποφάσεων για το πώς θα ολοκληρωθεί η ΟΝΕ και θα ήθελα να επισημάνω ότι όταν ε, θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση ε, στον κίνδυνο ασύμετρων κραδασμών πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτοί οι ασύμετροι κραδασμοί μπορούν οπωσδήποτε να μεταφραστούν ε, σε μια επιδείνωση της ανεργίας είναι σαφώς ένα κριτήριο αυτό αλλά μπορεί να μεταφραστούν και ως μια επιδείνωση της αξιολόγησης ε, της επενδυτικής, ειδικά της δημόσιας. Οπότε το μέσο το οποίο θα αναπτυχθεί θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη-μέλη στο να διατηρήσουν τις προσπάθειες για δημόσιες επενδύσεις, γιατί αυτό είναι σημαντικό για την οικονομική δυναμική, την ανάπτυξη και για να χρηματοδοτηθεί και η μετάβαση που πρέπει να χρηματοδοτήσουμε σε μια οικονομία έξυπνη και χαμηλό ανθρακά. Γι' αυτό ακριβώς ε, προτείνω μια τροπολογία που τα καλύπτει αυτά. Συνολικά όμως συμφωνώ με τις προτάσεις των εισηγητών και με τις τροπολογίες του κυρίου Σάντος για τον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ κυρία Ροντρίγκε. Θα δώσω τον λόγο και πάλι στον κύριο Λούκη μια που έχουμε λίγο χρόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο σημεία ήθελα να αναφέρω ακόμα. Το πρώτο αφορά την παρατήρηση του κυρίου Λάμπερτς, ο οποίος κατήγγειλε ότι κονδύλια του σχεδίου γιουνκερ Γιούνκερ-Ρέων κυρίως προς την Γερμανία και όχι προς χώρες που θα προτιμούσε ο ίδιος. Εδώ πέρα έχω να παρατηρήσω ότι ε, δεν είναι δυνατόν ε, να δώσουμε απλά λεφτά σε κάποιες ε, χώρες. Ο κύριος Ραμόν Τρεμόζα το ανέφερε. Είχαμε πάρα πολλές λανθασμένες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς πρώτης ευρωκρίσης, αυτοκινητόδρομους στους οποίους δεν ταξίδευε κανείς, ακίνητα τα οποία έμεναν άδεια και δεν απέδιδαν. Μία ουσιαστική αδυναμία της πρότασης αυτής της Κομισιόν είναι το ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται αυτομάτως ε, επενδύσεις χωρίς ε, να είναι κερδοφόρες. Δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος ε, κερδοφορίας. Όμως αυτή θα πρέπει να είναι η βασική προϋπόθεση οποιασδήποτε επένδυσης, ότι θα είναι αποτελεσματική, κερδοφόρα θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, απευθυνθήκα σε εσά και τώρα μια που έχουμε χρόνο στο πλαίσιο του KTI, εάν είναι δυνατόν οι δύο επιτροπές να δουν την νομική βάση. Τα άρθρα 174 και 175. σε τα επιχείρηματά μου για τα οποία θεωρώ ότι η Κομισιόν δρά εδώ πέρα ούλτρα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε εάν σκοπεύετε να ζητήσετε από την νομική υπηρεσία να εξετάσει την νομική βάση και το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Τώρα έχετε μιλήσει τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ δεν μπορώ να ε, εκφραστώ από πλευρά του κυρίου Γουαλτιέρη, αλλά θα στείλω το έτοιμά σα στην γραμματεία τη Επιτροπή Προπολογισμών. Ένα λεπτό, κύριε Φερνάντε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους συζητητές για την πρότασή τους, την, την οποία θεωρώ επικοδομητική και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς το νόμισμά μας, να ολοκληρωθεί λοιπόν η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Για το σχέδιο Juncker κυκλοφορούν ε, διάφοροι μύθοι και θρύλοι. Οι επενδύσεις πρέπει να δούμε πώς έχουν κατανεμηθεί όμως κατά χώρα και κατά οικονομία. Ποιοι επωφελήθηκαν περισσότερο με βάση και το ε, ΑΕΠ. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, μετά η Εστονία, μετά η Πορτογαλία. Αν τα συγκριβάλλουμε με βάση αυτά τα κριτήρια, αυτό θα διαπιστώσουμε. Όντω λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί ε, αυτό ο μηχανισμό και βοηθάει τα κράτη-μέλη που δεν μπορούν αλλιώ να κάνουν ε, επενδύσει. Και να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Τι είναι το InvestEU που είναι ένα πρόγραμμα που θα λειτουργήσει για την περίοδο 21-27, δεν μπορούμε να τον μπερδεύουμε λοιπόν με ένα μηχανισμό ε, χρηματοπιστωτικής ε, σταθεροποίησης ε, που είναι κάτι το οποίο θα παρεμβαίνει συγκεκριμένα, όχι συνεχώς, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες συγκυρίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες, λέει ο Οπότε, η συνεδρίαση ε, η συνεδρίασή μας η κοινή ε, θέλει να ακούσει τη γνώμη της Κομισιόν. Να την ακούσουμε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη θαυμάσια εργασία που έκαναν οι δύο επιτροπέ για να υποβάλουν αυτή την ιδιαίτερα επίκαιρη έκθεση και τροπολογίες ε, στην πρότασή μας για αυτό το μηχανισμό γίνεται μια συζήτηση που αποκτά όλη, όλο και περισσότερο στήριξη για έναν προπολογισμό της Ευρωζώνης και η πρότασή μας, όπως βελτιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση. Και ο μηχανισμός σταθεροποίησης, όπως ε, συζητείτε εδώ, μπορεί να είναι σημαντικός πυλώνας για τη διαμόρφωση του προπολογισμού της Ευρωζώνης, όπως προχωράει η συζήτηση και εξέταση αυτής της πρότασης. Εκτιμούμε λοιπόν τι προσπάθειε που έχουν γίνει. Δεύτερον, υπενθυμίζουμε ότι η πρότασή μα εστιάζει στην προσπάθεια ταχείας παρέμβασης για να ε, επιβραδυνθεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης χωρών που αντιμετωπίζουν ε, μια κρίση. Πρέπει λοιπόν να γίνεται γρήγορα η αποτίμηση των ε, επιλεξίμων επενδύσεων και να εκταμιεύονται ταχαίως οι πόροι για να παίξουν το ρόλο τους. Γι' αυτό στηρίζουμε τους εισηγητέ που ακριβώς τονίζουν ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να είναι απλά. Όσο πιο απλά γίνεται. Και σας καλούμε να αποφύγετε τον υπερβολικό ε, προκαταλογικό καθορισμό των επενδύσεων που θα είναι επιλέξιμες γιατί έτσι θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους χώρες που θα αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες ε, και ξαφνικές δυσχέρειες. Σημειώσαμε επίσης τη σαφή πρόθεση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού αυτού για να στηρίξει τα επιδόματα ανεργίας. Η Επιτροπή θα αναλάβει ιδιαίτερε πρωτοβουλίες εάν βεβαιωθεί αυτή η επιθυμία του Κοινοβουλίου και από τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν εκφράσει την, έκφραση, την στήριξή τους προς ε, αυτή την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Οπότε νομίζουμε ότι οι τροπολογίες που προτείνουν ε, οι συγητές είναι σωστή και βάσιμη τεχνική βάση για να ε, επεκτείνουμε λοιπόν και στη στήριξη των επιδομάτων ανεργίας την πρόταση αυτή. Πρόεδρος. Για να συνοψίσουν οι συνεισηγητές, ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, ο Μπέγκε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι για τις ε, παρεμβάσεις σας και για τα σχόλιά σας, τα θετικά σχόλια. Να παραθέσω δύο φράσεις από πρόταση σχετικά με την αρχιτεκτονική προπολογισμού της Ευρωζώνης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δημοσιεύθηκε από το Γάλλο και Γερμανό Υπουργό Οικονομικών σαν αφορά τη νομική βάση. Έχουν κάποια σχόλια από αυτού και λένε ότι η νομική βάση για τέτοιο μέσο θα μπορούσε να είναι το άρθρο 175 μαζί με το 182 και το 173 σε συνδυασμό με το 136. Εγώ είμαι απόλυτα υπέρ του να εξετάσουμε τη νομική βάση, αναμφισβήτητα χρειάζεται αυτό, να αποφευχθεί το επιχείρημα ότι είναι παράνομο αυτό που κάνουμε. Πρέπει να διευκρινιστεί η νομική βάση Υπάρχουν επαρκείς νομικές βάσεις. Στη συνθήκη της Ρώμης ήδη αναφερόταν υποστήριξη χωρών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Δεύτερον, στο τέλος λοιπόν οι δύο υπουργοί λέγουν ότι ο προπολογισμό της Ευρωζώνης θα πρέπει να ανήκει στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσης και το ύψος του προπολογισμού θα καθορίσει τους αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Τελεία. Υπάρχουν κάποια καλά σχόλια που αφορούν την ιδέα μας για την χρήση της ε, αρχής του, των εισοδημάτων που πρέπει να συμβάλλουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αλλά ο Γάλλος και ο Γερμανός Υπουργό Οικονομικών λένε ότι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφασίζουν για το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή είναι σαφή συνθήκη ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτήν την νομοθεσία το Συμβούλιο. Πρέπει να δούμε τη σωστή διατύπωση. Για να πετύχουμε υποστήριξη από την πλειοψηφία. Και θα πρέπει να υπάρχει πάντα και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Μπερές έχει το λόγο. Εγώ θα, αν μου επιτρέπετε, θέλω λίγο περισσότερο χρόνο πάνω σε αυτά που είπε και ο κ. Μπέγκερ, θα πρέπει να υπομειστεί τις ευθύνε του το Κοινοβούλιο. Ζήτησε πάντα αρμοδιότητα για τον προπολογισμό. Μιλάμε για προπολογισμό τη Ευρωζώνης και γι' αυτό συνεργάζονται οι δύο επιτροπές. Σε αυτή τη θητεία αυτό που θα ψηφίσουμε θα είναι το έμβριο της θέσεως του Κοινοβουλίου πρέπει να δούμε τι γίνεται και στο Συμβούλιο, σε αυτό υπόψη και τη συζήτηση Γαλλία και Γερμανία. Βλέποντα αυτά, πρέπει να δώσουμε μεγάλη εντολή, ισχυρή εντολή όσον αφορά ε, την νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Secret Μουραζά να πω ότι όσον αφορά τον ορισμό του ασύμετρου κλονισμού, εγώ δεν είμαι πανεπιστημιακή ούτε οικονομολόγος. Κάτι μου λέει ότι η συζήτηση αυτή ε, είναι καρποφόρα. Θα είναι καρποφόρα και μπορούμε να διεξάγουμε σεμινάρια πάνω σε αυτό. Ε, δεν επηρεάζει πάνω από το 1 τρίτο των κρατών μελών αυτός ο κλονισμός. Δεν ξέρω, όταν η Ελλάδα, η Ιταλία ή κάποια άλλη χώρα της Ευρωζώνης κλονιστεί, ε, αυτή έχει υποστεί το ασύμετρο σοκ. Αν το σύστημα ε, όμως το Ιταλικό ή κάποιο άλλο δεν επηρεάζεται μόνο η Ευρωζώνη. Ποιος είναι ο ορισμός του κλονισμού, του ασύμετρου. Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό τον ασύμετρο κλειδονισμό. Αν δεν αντιμετωπιστεί γίνεται μέσω επιμόλυνσης συμμετρικός κλονισμός ε, λόγω της σχέσης των οικονομιών μας. Το ξέρουμε αυτό. Σας ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο αναφερθήκατε στη φύση της συζητήσεως που στρέφεται γύρω από τη θέση που έχουμε με τον κύριο Μπέγκερ. Είναι αποδοτική προσέγγιση ε, πάνω σε αυτή μπορούμε να οικοδομήσουμε. Είπατε στην ομάδα διεξέγεται μια συζήτηση όσον αφορά την, ε, το επίδομα ανεργία, την αποζημίωση για την ανεργία. Με το Μπέργκε είχαμε την πρώτη έκθεση για τον προπολογισμό τη Ευρωζώνη και συμφωνούσαμε και σταματήσαμε ε, πάνω σε αυτό. Και εκεί ε, έχουμε την αντασφάλιση της ανεργίας, συμφώνησα και κάναμε τεράστιο βήμα και στην πρόταση βάλαμε πολλά στοιχεία κάτι παραπάνω από μια απλή ασφάλιση για την ανεργία. Ε, και αυτή είναι η βάση ενός συμβιβασμού. Ο κύριε Λούκε, σας απάντησε ο κύριος Μπεοκέ για την ε, νομική βάση. Να προσθέσω ότι αν δείτε τις εργασίες του Ζακ Ντελόρ, όταν μπαίναμε στο ευρώ, είπε ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να ειδωθεί λόγω του ευρώ ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συγκλήσεις ή αποκλήσεις στην Ευρωζώνη. Ποτέ δεν ακολουθήθηκε αυτό και έχουμε υποστεί ε, αυτό που ζούμε σήμερα, τις συνέπειες. Άρα ήρθε και ώρα να ε, εξετάσουμε το θέμα της συνοχής. Ένα λεπτό, ε, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι με κοιτάτε, παρά που δεν σας κοιτάω. Ευχαριστώ τον Ραμόν Τρεμόσα για την υποστήριξή του και να υποστηρίξω Αυτά που είπε ο Μάριο Ντράικ υποστήριξε ένθαρμα την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Φιλίπ Λαμπέρ που νομίζω ότι κατέριψε την αίθουσα και στον Κεντισόλ που τους ευχαριστώ για την ε, υποστήριξη της ε, αρχής που χρησιμοποίησαν στην προσέγγιση. Να πω ότι το 2014 η αποζημίωση του επίδομα ανεργίας που διανεμήθη εντός ευρωζώνης ήταν 200 δισεκατομμύρια ευρώ όταν προτείνουμε αυτό το ταμείο να πρικοδευτεί με 55 δισεκατομμύρια ε, ε, πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη το ρόλο που πρέπει να παίξει η λειτουργία αυτή της σταθεροποίησης. Τώρα για τις επενδύσεις που πρέπει να περιστρέφονται γύρω από το διακύβευμα του κλίματος υποστηρίζω την Πατσοευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή αλλά έχω την ίδια παρατήρηση όπως και το σχέδιο Juncker Α που τελικά δέχτηκαν ότι μπορούμε να έχουμε πιο θετικό προσανατολισμό όσον αφορά την ε, οικολογική, την, την μετάβαση ε, σε μέτρα για το κλίμα, αν υπάρχει σωστή υποστήριξη, μπορούμε να δούμε θετικά ε, την προσέγγιση των πρασίνων σε αυτό το θέμα. Και ευχαριστώ που με επιτρέψατε να ξεπεράσω κατά πολύ το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κυρία Μπερέζ, ολοκληρώθηκε το σημείο 4 τη ε, κοινή αυτή συνεδρίαση Μπατζέκον. Σημείο 5 είναι τα διάφορα, δεν υπάρχει κάτι στα διάφορα. Να σα υπενθυμίσω όμως ότι η συνεδρίαση των σχεδόν για που είχε πραγματιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σήμερα ανεβλήθη, ακυρώθηκε και θα λάβει χώρα 12 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, οπότε δεν θα γίνει ψηφοφορία στις 3 Δεκεμβρίου. Η επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου, εξακολουθεί να ισχύει αυτή η συνεδρίαση ε, στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και καλή όρεξη.